Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, ας περάσουμε στο τελευταίο σημείο της σημερινής ημερήσιας διάταξης, το υπαριθμό 10, να καλωσορίσω τον κύριο Βαντίμ Πριστάικο, Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας. Κύριε Πριστάικο, είναι πραγματικά μεγάλη τιμή που σας έχουμε εδώ μαζί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε τόσο γρήγορα την πρόσκλησή μας να απευθυνθείτε στα μέλη της Επιτροπής μας. Καλωσορίσατε πάλι στις Βρυξέλλες, μια πόλη που τη γνωρίζετε πολύ καλά καθότι ήσασταν επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ τελευταία δύο χρόνια μέχρι να διοριστείτε υπουργό Εξωτερικών της χώρας σας. Ο κύριος Πριστάικο έφτασε σχεδόν στην ώρα του, έτρεξε για να είναι εδώ μαζί μας, μόλις έφτασε από το Λουξεμβούργο που συμμετείχε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων η Ουκρανία συμπεριλήφθηκε στη μερίσια διάταξη, ενδεχομένω θα μπορούσε να μα δώσετε κάποιε πληροφορίε σε σχέση με τη συζήτηση αυτή. Φαντάζομαι ότι αναγνωρίζετε ορισμένου παλαιότερου ευρωβουλευτέ από διάφορε πολιτικέ ομάδε και συμφωνώ ότι και οι παλαιοί και οι θα πρέπει να προωθήσουμε μια στενή συνεργασία και να στενό διάλογο με την Ουκρανία, ένα πολύ σημαντικό εταίρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να τονίσω αυτή τη στιγμή πόσο έντονη και στενή είναι η συνεργασία μας με την Ουκρανία τα τελευταία χρόνια και σαφώς θα θέλουμε, να συνεχίσουμε τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια στον ίδιο δρόμο. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση σας δίνω κύριε Υπουργέ τον λόγο και δυνατόν θα ήθελα να μας πείτε περισσότερα πράγματα όσον αφορά το ευρωπαϊκό θεματολόγιο της κυβέρνησής σας. Ας αναφερθείτε δυνατόν στο ζήτημα της ασφάλειας, αλλά και σε πολλά άλλα ζητήματα τα οποία απασχολούν του συναδέλφου εδώ. Σα δίνω το λόγο λοιπόν για 15 λεπτά και κατά αυτόν τον τρόπο οι συνάδελφοι θα μπορέσουν εν συνεχεία να θέσουν και ερωτήσει. Μπορεί να ακολουθήσει μια ανταλλαγή απόψεων και κύριε Υπουργέ, πρέπει να σα πω ότι μεταδίδεται ζωντανά μέσω του διαδικτύου η συζήτηση αυτή. Έχετε λοιπόν το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας εδώ σήμερα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στην Επιτροπή σας. Εκτιμώ όλους ιδιαίτερο το ρόλο που δραματίζει η Επιτροπή σας, υποστηρίζοντάς μας με πολλούς και διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, ήσασταν παρόντες στις αποστολές παρακολούθησης των εκλογών μας δύο φορές το τελευταίο διάστημα και όσον αφορά τη συζήτηση με τους υπόλοιπους υπουργούς ε, εξωτερικών, ε, θα σας πω ένα πράγματα που είπα και σε αυτούς. Συζητήσαμε τρία βασικά ζητήματα. Πρώτον, το ζήτημα της ασφάλειας στην Ουκρανία. Η διαδικασία του Μίνσκα, ιδίως όσον αφορά την σύνθεση Νορμανδίας και τις σχετικές συζητήσεις. Πρώτον αυτό, δεύτερον, οι μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό της Ουκρανίας Ορισμένες φορές μας έχουν πει ότι δεν προχωρούμε αρκετά, άλλες φορές ότι πηγαίνουμε πολύ γρήγορα και το τρίτο ζήτημα που θίξαμε ήταν οι προσδοκίες μας, δηλαδή τι περιμένουμε εμείς από εσά, αλλά και τι περιμένετε εσείς από εμάς. Θα αναφερθώ στα τρία αυτά ζητήματα, θα ήθελα όμως να σας ευχαριστήσω πρώτα για την υποστήριξή σας, καθότι ε, συμβάλλετε πάρα πολύ στην ε, ανταλλαγή κρατουμένων. Ο κύριος Σέντσοφ ο οποίος απελευθερώθηκε και αυτός, κατάφερε να επιστρέψει στο σπίτι του λόγω της δικής σας υποστήριξης. Θεωρούμε ότι αυτή η ανταλλαγή κρατουμένων ήρθε την κατάλληλη στιγμή, δεν ήταν δίκαιη σε καμία περίπτωση, αλλά ήρθε την κατάλληλη στιγμή και θεωρώ ότι θα δώσει έναυσμα σε ένα δεύτερο κύμα, σε ένα δεύτερο γύρο ανταλλαγής κρατουμένων. Άνθρωποι οι οποίοι θα έπρεπε εδώ και πέντε χρόνια να είχαν απελευθερωθεί. Τώρα, πώ έχουν τα πράγματα στην Ουκρανία. Ορισμένα πράγματα τα γνωρίζετε ήδη, δεν πρέπει να τα επαναλάβω θεωρώ. Πρέπει να σας πω ωστόσο ότι βρισκόμαστε ακόμα σε ένα καθεστώς πολέμου με τη Ρωσία. Και έχουμε χιλιάδες άτομα τα οποία έχουν χάσει τη ζωή τους τα τελευταία χρόνια. Άνδρες, γυναίκες, στρατιώτες, αλλά και άμαχος πληθυσμός. Δεν θα σας δώσω τα αριθμητικά δεδομένα, τα γνωρίζετε πολύ καλά, ιδίω όσοι έρχεστε συχνά στην Ουκρανία, τα έχετε δει η διεισόμαση. Πρέπει να σας πω πάντως ότι στην Ουκρανία όλοι μας και ο πρόεδρος Ζελένσκι προσπαθούμε να καταβάλουμε σημαντικές προσπάθειες για να εφαρμόσουμε τις συμφωνίες του Μίνσκα στο βαθμό που μας το επιτρέπει όμως η συνεργασία με τη Ρωσία πάντα. Ελπίζουμε ότι τα πρώτα βήματα που ήταν κυρίως ανθρωπιστικής φύσης θα μας επιτρέψουν να γυρίσουμε σελίδα στις σχέσεις με τη Ρωσία. Τι έχουμε κάνει και αυτό ήταν προϋπόθεση σε σχέση με την συνεδρίαση τύπου Νορμανδίας. Η Ρωσία ήθελε δύο πράγματα να γίνουν πριν συναντηθούν οι ηγέτες με τη σύνθεση Νορμανδίας. Η τελευταία συνεδρίαση έγινε το 2016. Επομένως εδώ και τρία χρόνια δεν έχουν συνομιλήσει οι, οι, οι θέλουμε να προωθήσουμε περισσότερο την προσέγγιση Σταν Μάιερ. Θα σας έλεγα ότι κάθε ταξιτζήση ακόμα και κομωτής στην Ουκρανία γνωρίζει τι θα πει μέθοδος προσέγγισης Μάιερ. Δεν ξέρω αν ο ίδιος βέβαια ο πρόεδρος Μάιερ γνωρίζει τι είχε προτείνει τότε. Πάντως πρόκειται για μια πρόταση που έλαβε χώρα στο Βερολίνο κατά τη διάρκεια της γερμανικής προεδρίας. Μια πολύ σύντομη αν θέλετε προσέγγιση και μέθοδος, πολύ απλή που α, ελπίζω ότι θα εφαρμοστεί στην πράξη προβλέπει ένα ειδικό καθεστώς, ένα ειδικό νόμο που προβλέπεται για την περιοχή εκείνη που βρίσκεται υπό την κατοχή της Ρωσίας να μπορέσει σε επιχειρησιακό επίπεδο να αρχίσει να λειτουργεί η νέα αυτή νομοθεσία την πρώτη μέρα των τοπικών εκλογών. Ο νέος λοιπόν αυτός νόμος θα πρέπει να αποκτήσει μόνιμο καθεστώς όταν η ε, Υπηρεσία Παρακολούθησης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Δημοκρατικών Υποθέσεων του ΟΑΣΑ, του ΑΣΕ με συγχωρείτε, πει ότι ε, η κατάσταση έχει πλέον σταθεροποιηθεί. Νομίζω ότι ε, θα πρέπει εδώ να λάβουμε υπόψη μας καταρχάς την περιοχή στα Λουχάνσκα, όπου ήδη έχουμε αρχίσει να κατασκευάζουμε εκεί πέρα μια γέφυρα, η οποία σε μερικούς μήνες θα είναι έτοιμη. Επομένω, αυτό το έχουμε καλύψει. Υπάρχουν δύο ακόμα τομεί όμω που πρέπει να καλυφθούν. Περιμένουμε αυτή τη στιγμή να υπάρξει μία περίοδος παύσης του πυρός για 8 μέρες. Αυτό έχει αποφασιστεί και στο παρελθόν ότι μετά από μία επταήμερη τέτοια περίοδο παύσης του πυρός, την 8η μέρα, μπορούν οι δυνάμεις οι οποίες είναι στην περιοχή να αποχωρήσουν, να απεμπλακούν. Δεν έχει συμβεί αυτό ακόμα, αλλά ελπίζουμε ότι μέσα σε δύο εβδομάδες θα γίνει κάτι τέτοιο, πριν τα τέλη Οκτωβρίου δηλαδή. Και ελπίζουμε ότι κατά αυτόν τον τρόπο τους επόμενους μήνες θα μπορέσει να συνεδριάσει η τετράδα της Νορμανδίας. Αυτά όσον αφορά την ομάδα επαφής με τη σύνθεση της Νορμανδίας. Ξέρετε ότι η Ρωσία πολλές φορές εμφανίζεται προβάλλοντας συγκεκριμένες απαιτήσεις και προσδοκίες όσον αφορά στις συμφωνίες του Μίνσκ. Πάντως υπάρχουν συγκεκριμένες συμφωνίες του Μίνσκ, έχουν υποβληθεί αυτή τη στιγμή τρεις συγκεκριμένε απαιτήσει από τη Ρωσία και έχουμε καλύψει από κοινού τις δύο από αυτές. Έτσι έχουν τα πράγματα στην πράξη. Καταφέραμε να φέρουμε πίσω στην Ουκρανία 35 κρατουμένους. Θυμάστε ότι η κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη διότι η Ρωσία έπρεπε να ακολουθήσει εδώ πέρα μία απόφαση του δικαστηρίου. Έπρεπε να απελευθερωθούν και αυτοί οι 27 ναυτικοί πλήρωμα ουσιαστικά των σκαφών εκείνων που είχαν σταματήσει οι Ρώσοι στα στενά του Κέρτς. Προσπαθήσαμε επίσης να δούμε τι θα μπορούσε να γίνει με τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο έδαφος της Ουκρανίας. Έπρεπε να γίνει μια ανταλλαγή κρατουμένων, ακόμα και για τους κρατούμενους τρομοκράτες που είχαμε εμείς στην Ουκρανία, προκειμένου να καταφέρουμε να πάρουμε πίσω και να επαναπατρίσουμε τους ναυτικούς, αλλά και άλλους πολιτικούς κρατουμένους. Ελπίζουμε ότι η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί, προκειμένου να έχουμε το σύνολο των κρατουμένων πίσω στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι προσπαθεί να έρθει σε επαφή και με όσους βρίσκονται στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας Ελπίζουμε ότι εκεί πέρα θα μπορέσει να υπάρξει ένα καθεστώ, ένα μερικό καθεστώ αυτοδιάθεση, το οποίο θα περάσει ούτω ή άλλω από μία μέθοδο αποκέντρωση, η οποία ήδη έχει αρχίσει να εφαρμόζεται στην Ουκρανία. Υπάρχουν κάποιε κόκκινε γραμμέ, οι οποίε είναι πολύ απλέ. Η Ουκρανία είναι και θα παραμείνει ένα ενιαίο κράτο. Σε καμία περίπτωση δεν συζητάμε καμία ομοσπονδιοποίηση τη Ουκρανία. Δεύτερη κόκκινη γραμμή. Δεν πρόκειται να τροποποιήσουμε το Σύνταγμά μα με βάση τι προσταγέ τη Ρωσία. Μπορούμε και θα κάνουμε κάποιε μεταρρυθμίσει στο Σύνταγμά μα για να προωθήσουμε περισσότερο πολιτικές αποκέντρωση, όπως άλλωστε λέγεται και συμφωνίες Μίνσκα. Τρίτη κόκκινη γραμμή. Θα γίνουν εκλογέ προφανώ, αλλά οι εκλογέ αυτές θα διοργανωθούν βάσει του ουκρανικού δικαίου και βάσει των προτύπων του ΑΣΕ και όταν το επιτρέψει το κλίμα ασφάλειας αυτό. Δεν θέλουμε μισθοφόρους από τη Ρωσία, ούτε ρωσικά όπλα στο έδαφος της Ουκρανίας και θα πρέπει να αποσυρθούν τα ρωσικά στρατεύματα καθώς επίσης και οι αμυντικοί εξοπλισμοί της Ρωσίας. Διαφορετικά, αν δεν πληρωθούν, αν θέλετε, τα κριτήρια αυτά, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορέσουμε να έχουμε ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, καθότι θα βρίσκονται ουσιαστικά υπό την επιρροή της Ρωσίας. Ολοκληρώνω στο σημείο αυτό. Αν έχετε άλλες ερωτήσεις για την κατάσταση ασφαλείας στην Ουκρανία, μπορώ να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες. Όσον αφορά τώρα τις μεταρρυθμίσεις που έχουμε κάνει στην Ουκρανία, ξέρω ότι μας κατηγορούν μερικές φορές ότι έχουμε μια προσέγγιση ιδιαίτερα γραφειοκρατική ή ότι προσπαθούμε εντάχει να περάσουμε πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις. Ναι, αλλά το κάνουμε αυτό γιατί έχουμε χάσει πάρα πολύ χρόνο στο παρελθόν. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να εγκρίνουμε με τον συντομότερο δυνατό τρόπο πάρα πολλά νέα νομοσχέδια, τα οποία ούτω ή άλλω εκκρεμούσαν τελευταία πέντε, αν όχι και δέκα χρόνια. Ελπίζουμε λοιπόν ότι οι βουλευτέ μα θα καταφέρουν να, περά... να εξετάσουν αυτά τα 73 νομοσχέδια μέσα σε μερικού μόνο μήνε, σε ένα μήνα μάλλον. Καταλαβαίνετε ότι προφανώ θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια διαδικασία fast track. Δεν μπορούμε να κάνουμε ενδελεχή εξέταση όλων αυτών των νομοσχεδίων, αλλά μην ξεχνάμε ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να προωθήσουμε εντάχει αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Το επίτευγμα σίγουρα είναι, το διακύβευμα μάλλον είναι πολύ σημαντικό, αλλά έχει να κάνει με πολύ ευαίσθητους τομείς, όπως η καταπολέμηση της διαφθοράς, η μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, η μεταρρύθμιση του γραφείου του εισαγγελέα, στα ζητήματα αυτά καλούμεθα να πετύχουμε πολύ γρήγορα θετικά αποτελέσματα και προσπαθούμε ως νέα κυβέρνηση της Ουκρανίας να δείξουμε ότι όλα αυτά τα λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Τα πρώτα νομοσχέδια τα οποία φτάσανε στο Κοινοβούλιο μας είχαν να κάνουν με την ασυλία των βουλευτών. Ουσιαστικά θελήσαμε εδώ πέρα να λάβουμε κάποια δραστικά μέτρα για να καταπολεμήσουμε φαινόμενα διαφθοράς. Επίσης, συζητάμε αυτή τη στιγμή κάποιους βασικούς οικονομικούς νόμους που πρέπει να εγκρίνουμε το στομότερο δυνατό, καθότι ε, έχουν να κάνουν με τις υποχρεώσεις που έχουμε στο πλαίσιο της Συμφωνίας Σύνδεσης που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Πρόεδρος υπέγραψε μια συμφωνία πρόσφατα που μας ε, επιτρέπει να έχουμε ένα καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεωρήσεων, ιδίως στον βιομηχανικό επιχειρηματικό τομέα και μπορούμε αυτή τη στιγμή ουσιαστικά να προωθήσουμε πολύ περισσότερο την επιχειρηματικότητα στην χώρα μας. Σίγουρα έχουμε αναθεωρήσει πάρα πολύ τα συστήματα τοπικής αυτοδιοίκησης, Έχουμε αλλάξει την ηγεσία στις υπηρεσίες καταπολέμησης διαφθοράς ή ακόμα και την ηγεσία στις εισαγγελικέ μας αρχές και ελπίζουμε ότι όλα αυτά θα δώσουν πολύ γρήγορα επικοδομητικά αποτελέσματα. Και κάτι ακόμα. Να υπενθυμίσω ότι εμείς δεν έχουμε τροποποιήσει τον τρόπο με τον οποίο ατενίζουμε το μέλλον. Πιστεύουμε ακράδαντα στην ευρωπαϊκή μας προοπτική, στην προσχώρησή μας επίσης στο ΝΑΤΟ. Και αυτό δεν είναι μόνο μέρος πλέον του συντάγματός μας, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα βαθιά ριζωμένο στην ίδια την οτροπία πλέον και στη στάση που κρατούν οι ίδιοι οι πολίτες της Ουκρανίας και θεωρούμε ότι θα πρέπει να περπατήσουμε στο δρόμο αυτό της ευρωπαϊκής προοπτικής έχοντας και τη δική σας την υποστήριξη. Τη χρειαζόμαστε την υποστήριξη αυτή. Οι πολίτες της Ουκρανίας την χρειάζονται, τη βοήθειά σας και τη δική σας συνδρομή στον καθημερινό αγώνα το οποίο δίνουν. Ολοκληρώνω σε αυτό το σημείο κύριε Πρόεδρε και προσβλέπω σε ερωτήσεις των συναδέλφων σας. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Να δώσω πρώτα τον λόγο στον επικεφαλής ε, της Αντιπροσωπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με την Ουκρανία που είναι και αντιπρόεδρος της Επιτροπής μας, τον κύριο Βασικόφσκι. Ευχαριστώ, σας καλωσορίζω και εγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως είπε ο Πρόεδρος, εγώ θα είμαι Πρόεδρος της ε, Αντιπροσωπείας ε, Κοινοβουλευτικής για τις σχέσεις μεταξύ του δικού μας Κοινοβουλίου και του Κοινοβουλίου της ε, Ουκρανίας και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα εκλεγεί και η ομόλογη αντιπροσωπεία της ΡΑΝΤΑ και θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη δουλειά που μας περιμένει τα επόμενα λίγα χρόνια. Πρέπει να γνωριστούμε όχι βεβαίως από την αρχή, γιατί υπάρχουν κάποιοι βετεράνοι και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην, ε, στο Κοινοβούλιο της Ουκρανίας. Ξέρω όμως ότι περίπου το 80% των βουλευτών ε, στο Κοινοβούλιο της ε, Ουκρανίας είναι νεοεκλεγέντε. Ε, αντίστοιχα, λιγότερο βεβαίω, αλλά αντίστοιχα υπάρχουν και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολλοί νέοι ευρωβουλευτέ, οπότε πρέπει σχεδόν από την αρχή να ξαναγνωριστούμε θα επιχειρήσω εγώ βεβαίως να επικεντρώσουμε την δουλειά μας ε, στην εμβάθυνση του πολιτικού διαλόγου μεταξύ των θεσμικών οργάνων μας με προγράμματα καλής διακυβέρνησης για παράδειγμα ή που αφορούν το κράτος δικαίου. Γιατί με την εφαρμογή αυτών ε, θα, ωφελευ... θα ωφεληθείτε και από την οικονομική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως δεν μπορώ να ξεχάσω τα προβλήματα ε, της ασφάλειας ε, που αντιμετωπίζει η Ουκρανία είστε γείτονας της ε, Πολωνίας, είστε γείτονας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την άλλη μεριά έχετε έναν γείτονα, τη Ρωσία, που επιδεικνύει μεγάλη επιθετικότητα και εσείς είστε το θύμα της επιθετικότητας αυτής. Θέλω λοιπόν να σας διαβεβαιώσω ότι τα ζητήματα της ε, εδαφικής ακαιρεότητας και της ασφάλειας της Ουκρανίας θα παραμείνουν πολύ ψηλά στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφοι, έχουμε περίπου μισή ώρα στη διάθεσή μας. Έχω δέκα συναδέλφους που μου έχουν ζητήσει το λόγο. Να διαβάσω τα ονόματα. E για το ΕΛΚ, για το σοσιαλιστές, for Renew Ostrevichus, Renew πράσινος, η κυρία Καπτομτόμπ Άμπελ, η κυρία Φωτίκα για το ECR, ο κύριος Γόλης για την ΚΟΕ και από τους μη εγγεγραμμένους ο κύριος Παπαδάκης και ο κύριος Κουμπίλιος. Ωραία, να του ακούσουμε όλους. Πολύ ωραία. Δύο λεπτά, αν μπορείτε, σας παρακαλώ. Ο κύριος Μιχαήλ Γκάλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ ε, που εξηγήσατε αυτή τη φόρμουλα Steinmeier και συμφωνώ επίση και με, το, με αυτά που είπατε όσον αφορά την αλληλουχία των όσων πρέπει να γίνουν σε περίπτωση που εφαρμοστεί. Είναι η μόνη λογική, αν θέλουμε κάποια στιγμή να φτάσουμε σε εκλογέ. Όλα αυτά τα ζητήματα που αναφέρατε πραγματικά πρέπει να προηγηθούν. Τώρα, κάποια ερωτήματα σχετικά με συγκεκριμένα βήματα ε, των μεταρρυθμίσεων. Τι, πώς προχωράει η αποκέντρωση και τι σχεδιάζεται για την ε, ολοκλήρωση της αποκέντρωσης. Για το ε, δικαστήριο κατά της ε, και τα έγγραφα της ΝΑΜΠΟΥ. Αυτά τα έγγραφα δεν θα έπρεπε να είχαν φτάσει στο σύστημα εκεί, αλλά τελικά ε, έγινε αυτό. Πώς μπορεί λοιπόν η ΝΑΜΠΟΥ να συντάξει αυτά τα έγγραφα και να τα αφήσει στο, και να τα παραδώσει στον ΝΑΚ. Επίσης, Στι συνδιάσκεψη ΓΕΣ ε, υπάρχουν πολλά ερωτήματα σε σχέση, με τον κύριο ε, Χοροσόφσκι, τον οποίο εγώ τον είχα, ε, τον είχα συναντήσει ε, την εποχή Γιαννούκοβιτς, ε, που έκανε και αυτός μια επανεμφάνιση. Είναι ανάγκη να εμφανίζονται αυτοί οι άνθρωποι δίπλα στη νέα κυβέρνηση. Τέλος, μεταρρύθμιση του συστήματος υγείου, υγείας. Έχουμε την εντύπωση ότι ε, υπάρχουν κάποια κέντρα τα οποία θέλουν οι οικονομικές ροές, οι ροές των χρημάτων να, να κατευθυνθούν αλλού από ό,τι προβλέπει ο νόμος. Ο κύριος Πίτσουλα. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου η Ουκρανία πάντοτε βεβαίως ε, ε, έχει πολύ μεγάλη υποστήριξη. Τρία θέματα θέλω να θέσω. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι Ευρωβουλευτέ ε, παρακολουθούν στενά την ε, πρόοδο που σημειώνει η Ουκρανία στι μεταρρυθμίσει, ιδίω τη δικαιοσύνη και το έργο των νέων οργάνων και φορέων για την καταπολέμηση τη διαφθοράς. Γι' αυτό και σα ε, ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιήσετε όλε τι δυνατότητε παροχή συμβουλών από εμά για το πώ μπορείτε να προετοιμαστείτε για την, για την εφαρμογή μια τέτοια σημαντική μεταρρύθμιση, για παράδειγμα αξιοποιώντα ε, την εμπειρογνωμοσύνη της Επιτροπής της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Θα ήθελα ε, να μου πείτε κι εσείς ποια θα είναι τα επόμενα βήματα που σχεδιάζετε στη μεταρρύθμιση δικαιοσύνης. Δεύτερον, ε, θέλουμε να υποστηρίξουμε την ε, προσπάθεια που γίνεται για την επίλυση των προβλημάτων της ε, Ανατολικής Ουκρανίας και την νέα διαδικασία της Νορμανδίας, εκφράζοντας ταυτόχρονα την υποστήριξή μας στην εδαφική ε, ε, ακαιρεότητα της Ουκρανίας. Η, επίσης, έχουν εκφραστεί συγκεκριμένε εκτιμήσει όσον αφορά τι χρηματοδοτικέ ανάγκε που θα έχει η ανακοδόμηση του Ντομπά. Ποιε είναι οι δικέ σα εκτιμήσει, Επίση, ε, υπάρχει μια κρίση εμπιστοσύνης ε, στο Συμβούλιο της Ευρώπης έπειτα από την επιστροφή της αντιπροσωπείας της Ρωσίας. Πώς βλέπετε εσείς ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε, αυτήν, την, ε, σε αυτόν τον τομέα. Ευχαριστώ για το ε, Renew, ο κύριος Οστρεβίτσιος. Ευχαριστώ. Σας καλωσορίζω κύριε Υπουργέ. Μόλις επέστρεψα από το Λονδίνο, όπου είχαμε μια εξαίρετη σύνοδο ε, όπου συζητήσαμε πολύ ε, πισταμένα την κατάσταση στην Ουκρανία και τα συμπεράσματα είναι πολύ ε, σταθερά και γι' αυτό θα πρέπει να επιμείνουμε για να έχουμε περισσότερη υποστήριξη για την Ουκρανία για το επόμενο διάστημα. Εκτιμούμε ε, ιδιαίτερα τώρα ε, τις μεταρρυθμίσεις του Προέδρου ε, Ζαλένσκι, εμείς, και ε, όμως η κοινή γνώμη τι λέει. Ε, όσον αφορά τις πιθανές ειρνευτικές διαπραγματεύσεις ε, Πόσο μπορεί λοιπόν να στηριχτείτε ε, στην ε, δημόσια υποστήριξη έπειτα και επεκτηνόμενος με βάση την ερώτηση του κ. Πίτσουλα, τι, μπορείτε, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια για το τόμπας, για να ε, υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες να βοηθήσουμε, αλλά και δέσμευση του Κίεβου ώστε να θα δώσουμε στον κόσμο μια πιο θετική εικόνα για ένα μέλλον, να μην τους αφήσουμε σε αυτή την ρωσική προπαγάνδα και την επιρροή της Μόσχας. Έπειτα υπάρχουν ε, νέα ή καλά νέα για το τι συζητήθηκε μεταξύ του Προέδρου Ζαλένσκι και του Προέδρου Λουκασέγκο γιατί υπάρχει, γίνεται, ακούγονται διάφορα για την Λευκορωσία, για ανεξαρτησία υποτιθέμενη της Λευκορωσίας. Εσείς πώς βλέπετε την κατάσταση με το βόρειο σας γείτονα. Ευχαριστώ πολύ. Πέτρα Σωστοβίτσιος από τους Πράσινους. Η κυρία Κράμον Τόμποντελα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επειδή είμαι και αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας, θα ήθελα να τονίσω αυτό που είπε ο επικεφαλή της Αντιπροσωπείας μας, ότι ναι, ε, ενδιαφερόμαστε πολύ στο να ξεκινήσουμε και να συνεχίσουμε εντατικό διάλογο με τους βουλευτές και βλέπουμε ότι υπάρχει τέτοια βούληση από το Ουκρανικό Κοινοβούλιο αλλά και από εμά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, ιδιαίτερα όσον αφορά την κατάσταση στην Ανατολική Ουκρανία, την ασφάλεια, θα ήθελα να, πείτε, να μου πείτε γιατί, τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα, για την ανταλλαγή κρατουμένων που είπατε, εσείς δώσατε πολλά και πετύχατε κάτι, αλλά υπάρχει ασυμμετρική κατάσταση. Μπορείτε να φανταστείτε τι, ποιο θα είναι το επόμενο βήμα ε, υπό τη μορφή του Μίνσκ ή της Νορμανδίας. Η Μόσχα θα δεχτεί αυτό που εσείς ζητήσατε, το ποια θα είναι δηλαδή τα επόμενα βήματα. Εγώ δεν καταλαβαίνω πραγματικά πώς θέλετε να χειριστείτε αυτές τις εκλογές, ποιος θα τις υποπτεύσει. γιατί εντάξει εμεί θα μπορούμε να έρθουμε σαν παρατηρητέ, αλλά από την Ουκρανική πλευρά ποιο θα είναι υπεύθυνο, είναι υποσυζήτηση η αποστολή τη Ένωση και τι είδου διεθνή εποπτεία ε, θα ε, θα κάνει τον ε, επιτήρηση. Δεν ξέρω κατά πόσο θα δεχτεί των, ε, εκεί τις διαφανείς ε, και ανεξάρτητες αδιάβλητες εκλογές. Για μας δεν υπάρχει σαφής γραμμή. Ο Γερμέκο είναι περισσότερο σκιαώδης για τον Υπουργό ή για το ποιος είναι επικεφαλής για αυτή την ε, φόρμουλα, για αυτή τη συμφωνία. Μπορείτε κάποια περισσότερα πράγματα να μας πείτε. Ποιος θα ηγηθεί αυτών των διαπραγματεύσεων. Και πραγματικά δεν θα πρέπει να αναμειχθεί η διαδικασία αποκέντρωση στην Ουκρανία με τη φόρμουλα του Μίνσκ. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος του ECR η Άννα Φωτίγα. Καλώς ορίσατε, Υπουργέ, στην ΑΦΕΤΑ. Συνεχίζει η υποστήριξη η στεναρή μας προς την Ουκρανία όσον αφορά την εδεφική της ακυριότητα και την αντίσταση στη ρωσική ε, βία. Έχω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, ποια είναι η δική σας εκτίμηση για την ελευθερία πλοήγηση στη θάλασσα Ζόφ και τα στενά του Κέρτς και έπειτα ποια είναι η τουρκική θέση για την, τουρκική, για την ακαιρεότητα της Ουκρανίας. Okay, thank you, Anna. For the GUI group, Mr. Wallace. Wallace από την GUE. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για την εισήγησή σας. Ο Σαλένσκι κέρδισε μεγάλη υποστήριξη, 72% στις εκλογές και ε, ήθελε και μάλιστα βασίστηκε στην υποστήριξη της ειρήνης. Είναι σαφές πως ο λαός της Ουκρανίας θέλει την ειρήνη. Ο μόνος που ενδιαφέρεται λιγότερο είναι κάποιες νεοναζιστικές ομάδες καθώς και εκείνοι που κερδίζουν από την πώληση όπλων. Και μιλώντας για όπλα, η Ουκρανία, όπως είμαι βέβαιος γνωρίζετε καλύτερα από μένα, αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις. Διαρωτώ με γιατί μια χώρα να δαπανά τόσα χρήματα στα όπλα ενώ έχει να αντιμετωπίσει τόσες άλλες προκλήσεις. Διότι αυτό δεν πρόκειται να ε, ε, σας βοηθήσει στο να χορτάσει ο λαός σας. Τώρα, ε, Αναφέρθηκε και η ιδιωτικοποίηση και γνωρίζουμε πως όταν η Ρωσία ξεκίνησε την ιδιωτικοποιήσει τις ιδιωτικοποίησεις υπό τον Γέλτζεν, αυτό αύξησε τη διαφθορά. Οι μόνοι που ωφελήθηκαν ήταν οι ολιγάρχες. Αληθεύει ότι ο Ζελένσκι σκέφτεται να ιδιωτικοποιήσει μεγάλα κομμάτια γης που είναι κρατική περιουσία για την ώρα. Επίσης, Μπορείτε να μου πείτε γιατί συνάντησε την νεοναζιστική ή E14 πριν από λίγες μέρες. Αναγνωρίζεται ως τρομοκρατική οργάνωση ε, ε, εκεί αναζήτησε μήπως τη στήριξη των νεοναζί στην ειρηνευτική διαδικασία και έπειτα ε, χτες ο Πρωθυπουργός Χάνσροφ παρακολούθησε μια συναυλία βετεράνων ε, που διοργάνωσε πάλι η 14. Για ποιο λόγο λοιπόν παρακολούθησε, ε, εκεί, πήγε εκεί μάλλον ο Πρωθυπουργό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παπαδάκης. Δύο λεπτά. I will speak in Greek. Uh, Κύριε Υπουργέ, στις 16 του Ιούλη το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ουκρανίας επέβαλε την απαγόρευση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ουκρανίας. Στις 19 Αυγούστου απαγορεύτηκε από το Διοικητικό Δικαστήριο του Κιέβου η κυκλοφορία της εφημερίδας «Ραμπότσα για Γκαζέτα» του Κομμουνιστικού Κόμματος Ουκρανίας. Επίσης, του απαγορεύτηκε και το δικαίωμα να κατέβει στις εκλογές. Τα παραπάνω αποδεικνύουν τα υποκριτικά συνθήματά σας περί ελευθερίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικών ελευθεριών. Η κυβέρνησή σας, όπως και οι προηγούμενες, κάνουν τις πλάτες εφασιστικές συμμορίες και είναι αλήθεια όσα υπόθηκαν από τον προηγούμενο συνάδελφο, συμμετέχει και τιμά απόγονους των Ναζί και προκλητικά και ανιστόρητα με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξισώνει τον κομμουνισμό με το τέρας του φασισμού. Τι έχετε να πείτε λοιπόν απέναντι σε αυτές τις απαράδεκτες και εξοργιστικέ αποφάσει και στο αναφέρετο δικαίωμα στην πολιτική δραστηριότητα των κομμουνιστών στην ανεμπόδιστη διάδοση των ιδεών του. Ευχαριστώ. Thank you. And now we finally come to an... E- Ευχαριστούμε πολύ. Α ακούσουμε τώρα ρωτήσεις από το ΕΛΚΑ. Η κυρία Κανιέτη πρώτη. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζουμε στην Επιτροπή μας. Καταρχάς, όσον αφορά την προσέγγιση Μάιερ, χάρηκα πάρα πολύ που αναφερθήκατε στις κόκκινες γραμμές που είναι πάρα πολύ σημαντικές για την Ουκρανία. Από την άλλη όμως, καθότι γνωρίζω πολύ καλά την πολιτική που ακολουθεί η Ρωσία και τα εργαλεία τα οποία έχει, όπως για παράδειγμα η διεθνής της προπαγάνδα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην γίνετε εσείς οι ένοχοι όσον αφορά τη διεθνή κοινότητα γιατί η Ρωσία μετά από λίγο θα αρχίσει να σας κατηγορεί για έλλειψη επιτυχίας και έλλειψη πολιτικής βούλησης όσον αφορά την εφαρμογή της φόρμουλας Μάιερ. Στο παρελθόν, όταν οι βαλτικές χώρες κέρδισαν την ανεξαρτησία τους, δεν ήταν 70% αλλά 95% το ποσοστό των ε, βουλευτών που πρώτη φορά εκλεγόντουσαν και βλέπετε που έχουμε φτάσει σήμερα. Πολλές φορές αυτό είναι πλεονέκτημα, να μπορεί να μάθει κανείς από τις καλές και όχι τις κακές πηγές. Και δύο ερωτήσεις. Πρώτον, η σύνδεση αυτή που υπάρχει μεταξύ της Τράπεζας Πρίβεν και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. και η εκταμείευση των κονδυλίων για την Ουκρανία. Αναφέρομαι εδώ πέρα στην απενεθνικοποίηση της τράπεζας αυτής. Θα ήθελα σωστικά να γνωρίζω πώς θα εφαρμοστεί καταρχάς η νομοθεσία όσον αφορά την γεωργική μεταρρύθμιση και τη μεταρρύθμιση της ιδιοκτησίας των γεών. Η Ουκρανία έχει, ε, έχει από τις πιο έφορες γεωργικές εκτάσεις στην Ευρώπη. Οπότε καταλαβαίνετε πόσοι πολλοί θα είναι οι επενδυτές οι οποίοι ε, ήδη από τώρα σκέφτονται ότι θα μπορούσαν να αποκτήσουν ε, αγροτεμάχια από την Ουκρανία. Ακριβώς αυτό γνωρίσαμε και σε βαλτικές χώρες, αλλά και σε χώρες όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία διότι το πρόβλημα είναι ότι συνήθως οι επενδυτές απ' έξω έχουν πολύ περισσότερα χρήματα. Διακαώς θέλουν να αγοράσουν τις εκτάσεις σας και εσείς θα πρέπει τρόπον την να τις προστατεύσετε. Θα ήταν πολύ σημαντικό λοιπόν να μας δώσετε μια σφαιρική εικόνα των πραγμάτων και από αυτού περιμένω και τα σχόλιά σας. Ευχαριστούμε ο κύριος Μπαζέσκου τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Νομίζω ότι εδώ, αν θέλετε, ο κατάλληλο χώρος για να συζητήσουμε την κατάσταση της Ουκρανίας. Δύο ερωτήσει θα ήθελα να κάνω. Πρώτον, θα είμαι πολύ ειλικρινής, πραγματικά μου έκανε εντύπωση ο τόσο εύκολος τρόπος με τον οποίο εγκρίθηκε η προσέγγιση Μάιερ από την Ουκρανία. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι αναφερόμαστε εδώ πέρα σε ένα είδος υπευνηστερίας, αν θέλετε, για την Ουκρανία, ότι ένα ανάλογο καθεστώς αυτή τη στιγμή θα αρχίσει να ισχύει σε περιοχές όπως το Λουγκάνσκ ή το Ντον Δεν Μπορούμε να λέμε ότι η Ουκρανία θα είναι ένα ενιαίο κράτος τη στιγμή που διακυβεύονται τόσο σημαντικά ζητήματα. Από ό,τι φαίνεται θα είναι τεράστιες οι εκτάσεις αυτές οι οποίες θα ενταχθούν στην νέα αυτή διοικητική διάρθρωση που προβλέπεται. Και βλέπετε ότι η Ρωσία κατάφερε προωθώντας τις δικές της διεκδικήσεις να πετύχει, θα πετύχει αν εφαρμοστεί η πρόταση αυτή κατά 100% να περάσει στη δική της ιδιοκτησία τα εδάφια αυτά. Όσον αφορά το άρθρο 4 τώρα, τη Συμφωνία Σύνδεσης που έχετε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια συμφωνία που έχω υπογράψει και εγώ ο ίδιος πρέπει να σας πω, Εκεί γίνεται αναφορά στις μειονότητες. Βέβαια, εγώ δεν μπορώ να κρίνω ή να επικρίνω την κυβέρνηση, το κοινοβούλιο της Ουκρανίας, αλλά κατά την άποψή μου έχετε κάνει ένα σημαντικό λάθος εδώ. Όταν αποφασίσατε να μην επιτρέψετε στις μειονότητες να μπορούν να χρησιμοποιούν και να μαθαίνουν την εθνική τους γλώσσα, για παράδειγμα την ουγγρική ή την ρουμανική γλώσσα. Και ανταυτού υποχρεώνεται τις μειονότητες αυτές να εκπαιδεύονται στην ε, ουκρανική μόνο γλώσσα. Καταλαβαίνετε το ζήτημα αυτό μπορεί να προκαλεί συντάσεις και στο δυτικό τμήμα της Ουκρανίας. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπαζέσκου, πρώτη τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Μπότσκο. Um, ευχαριστώ και σας ευχαριστώ που ήρθατε κύριε Υπουργέ. Τα ερωτήματά μου συνδέονται με ορισμένα από τα ερωτήματα που έθεσαν ήδη κάποιοι άλλοι συνάδελφοι ή σχόλια που έκαναν. Πρώτο ερώτημα. Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια σχετικά με τις εθνικές μειονότητες. Γιατί ο πρόεδρος Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι θα Υποβάλλει ξεχωριστό νομοσχέδιο για το ζήτημα των εθνικών μειονοτήτων. Ε, τι θα περιλαμβάνει αυτό το νομοσχέδιο. Έχουμε κάποιες πληροφορίες από τώρα. Θα μπορούσατε να μας δώσετε κάτι. Δεύτερο ερώτημα σχετικά με τη διοικητική μεταρρύθμιση. Κυκλοφορούν φήμες ότι η Τρανσκαπάσια θα ε, συνδεθεί με το όμπλας του Λιβύβ. Είναι φήμες ή υπάρχουν και ψήγματα αλήθειας σε, αυτή, σε αυτές τις φήμες. Και τρίτο ερώτημα. Ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του Υπουργού Εξωτερικού όσον αφορά την έγκριση διπλωματικών σχέσεων με ε, γειτονικές ε, της Ουκρανίας χώρες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το ερώτημα. Ευχαριστώ. Και Τέλος, ε, ο κύριος Κομπίλου, πρόεδρος ε, της κοινοβουλευτική Συνέλευσης Euronest. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Δύο ερωτήματα. Η ειρηνευτική διαδικασία πρώτον. Μόνο να συγχαρούμε μπορούμε την Ουκρανική ηγεσία για, το, για την στάση της, αν και το κλειδί της ειρήνης βεβαίως βρίσκεται στο Κρεμλίνο και όχι στο Κίεβο. Αλλά βεβαίω δεν μπορούμε να αναγκάσουμε και την Ουκρανική ηγεσία να ε, ακολουθήσει ένα πρόγραμμα μη ρεαλιστικό. Είπατε λοιπόν ότι θα γίνουν εκλογέ στο Ντόνμπα. Ε, ε, βάσατε, βάλατε κάποια κριτήρια, όχι παρουσία μισθοφόρων κτλ. Που είναι απολύτω σωστά κατά τη γνώμη μου. Θα, θα είστε σε θέση να επιτύχετε αυτές τις προϋποθέσεις έως το τέλος ε, της επόμενης χρονιάς. Όχι φέτος, του 2020. Γιατί ξέρω ότι έχετε τοπικές εκλογές κάποια στιγμή το 2020. Και αν όχι, εσείς είπατε ανοιχτά για κάποιο σχέδιο Β που έχετε, δεν θυμάμαι τώρα πώς ακριβώς το αποκαλέσατε, σχετικά με το πάγωμα της ε, σύγκρουσης ή το να ακολουθήσετε ίσως το μοντέλο της Κύπρου. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο περισσότερο τι εννοείτε με αυτό. για την ειρηνευτική διαδικασία. Πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι η ειρήνη αυτή τη στιγμή δεν εξαρτάται μόνο από την Ουκρανία. Και αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερε γεωπολιτικέ προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ήπορο, Ήπειρο αυτή τη στιγμή. Πιο περίπλοκη και από τον Brexit. Κατά τη Σύνοδο Ολομέλεια εδώ στι Βρυξέλλε, εγώ πρότεινα να δημιουργήσουμε, αφού ε, είπα ότι αφού έχουμε ειδική διευθύνουσα επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Brexit, γιατί δεν έχουμε μια αντίστοιχη και για την Ουκρανία. Στην οποία θα μπορούσατε και εσείς βεβαίως να συμβάλλετε και να τροφοδοτείτε τις συζητήσεις μιας τέτοιας επιτροπής. Αυτά και σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, ήταν ευρύτατο το φάσμα των ερωτημάτων που ακούσατε. Είδατε ότι η Ουκρανία έχει πάρα πολλούς φίλους εδώ στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Πολλοί φίλοι παρακολουθούν εδώ και πολλά χρόνια την κατάσταση τη χώρα σα ενδιαφέρονται πολύ και είναι πλέον η ευκαιρία σας σε 15 λεπτά να απαντήσετε σε όλα αυτά τα ερωτήματα που ακούστηκαν. Ε, ανησυχώ, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ. Πάντοτε θαυμάζω την ικανότητά σας να συνθέτετε απόψει. Εγώ θα καλύψω τα περισσότερα από τα ζητήματα που σχετίστηκαν, αλλά θέλω να σταθώ στους ε, ε, ναζιστές, στους κομμουνιστές, στο Σιφουτίν και στο πώς μπορούμε να ξοδεύουμε χρήματα για όπλα όταν δεν έχουμε να φάμε. Δεν είναι ότι δεν έχουμε και να φάμε, κάτι τρώμε κι εμεί στην Ουκρανία. Με τη δική σας βοήθεια από το 0 μέσα σε 5 χρόνια καταφέραμε να φτάσουμε σε ρυθμό ανάπτυξη 4,6%. Αυτό δεν θα μπορούσαμε να το είχαμε καταφέρει χωρίς την πολιτική και οικονομική υποστήριξη των φίλων και συναδέλφων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μας βοήθησαν να στήσουμε την οικονομία μας στα πόδια μας. Τώρα μπορούμε ε, να συμβάλλουμε και εμείς λίγο στον ε, σχεδιασμό για το πώς θα βγούμε από αυτή τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρεθήκαμε. Το αν θα ξοδέψουμε τα χρήματα σε όπλα ή αλλού, εγώ καταρχά δεν συμφωνώ με την εκτίμησή σας. 2,3% είναι ο προπολογισμό μας για την άμυνα, που είναι το όριο ε, του ΝΑΤΟ για χώρες που δεν ε, βρίσκονται σε πόλεμο για την άμυνα και την ασφάλεια. Εγώ πιστεύω ότι 30% θα έπρεπε να ξοδεύουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την επιθετικότητα εναντίον μας. Ωστόσο, φυσικά ο μικρός κόκκινο στρατός δεν μπορεί να ε, νικήσει τον μεγάλο κόκκινο στρατό, οπότε για να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας αποτελεσματικά ε, χρειαζόμαστε και ε, χερσαίες ένοπλες δυνάμεις και αεροπορία και ναυτικό πολεμικό ναυτικό. Ξέρετε ότι ε, έχουμε μόλις ένα πολεμικό πλοίο. Όλα τα άλλα μας τα πήρε η Ρουσία. Και μάλιστα το πλοίο αυτό βρισκόταν σε αποστολή του ΝΑΤΟ. Ευτυχώς, χάρη στο ΝΑΤΟ δηλαδή, μας έμεινε και αυτό το ένα πολιτικό πολεμικό ε, πλοίο. Για τους νεοναζί και το έθνος είναι πολύ δύσκολο βεβαίως, ξέρετε, να κατηγορήσετε έναν Εβραίο του Νότου της Ουκρανίας, όπως είναι ο, κύριος ε, Ζελένσκι, ότι είναι ναζιστής. Ξέρετε ότι έχουμε, είμαστε η μόνη χώρα που είχαμε πρωθυπουργό και πρόεδρο Εβραίους ταυτόχρονα ε, και προφανώς δεν μπορούν ε, αυτοί οι άνθρωποι να κατηγορηθούν ως νεοναζί. Το να προσπαθεί κανείς να κατηγορήσει τους Ουκρανούς ως νεοναζί, τι, τι, να σας πω, όταν ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο ε, θυμάμαι ότι κάποιοι μα, μας έθεσαν το ζήτημα ναι υπάρχουν όμως και κάποιοι ε, εξτρεμιστές. Ναι, ε, απαντούσαμε. Χρειάζεται, αναγκαζόμαστε να αξιοποιούμε και τους εξτρεμιστές όταν ε, χάνουμε κόσμο, όταν σκοτώνεται κόσμο στο έδαφος μας, όταν ε, μπαίνει η Ρωσία και μας παίρνει μια ολόκληρη χερσόνησο. Όταν η ίδια η η, Ρωσία ε, ε, ε, γεμίζει τα εδάφη μας με νάρκες, βομβαρδίζει. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά για την οικονομία και τη βιομηχανία της Ουκρανίας. Ναι, εθνικά υπήρξε μια ριζοσπαστικοποίηση. Όμως πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι οι Ουκρανοί θα επανέλθουν στον δρόμο της κανονικότητας, στον συνήθι δρόμο, σε, αυτόν τον, σε, αυτόν τον, σε αυτή την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε ε, πάντοτε ε, ενός φιλήσυχου ε, αγροτικού λαού. Ε, αυτό όμως θα το καταφέρουμε όταν μόνο εφόσον με πειθαρχία όλες οι ομάδες υπό, υπό τον έλεγχο της κεντρικής Ουκρανικής κυβέρνησης αγωνιστούν για τον στόχο που έχουμε θέσει. Ε, αυτό είναι το, ο στόχος. Ε, αν δείτε σήμερα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, υπάρχουν διαμαρτυρίες και διδηλώσεις και μάλιστα μαζικές στους δρόμους της Ουκρανίας και προσπαθούμε να συνέλθουμε, να, να έρθουμε και σε επαφή με ομάδες οι οποίες μας λένε ότι η φόρμουλα Steinmeier είναι είναι συνθηκολόγηση. Εμείς ε, ε, δεν είμαστε τόσο αφελείς. Ξέρουμε, και εγώ ως διπλωμάτης δεν πιστεύω σε τίποτα, αλλά υπάρχουν ακόμη και ε, άνθρωποι ε, μέσα στην κυβέρνηση, γιατί ξέρουμε ότι η Ρωσία αν ήθελε και πριν από πέντε χρόνια θα μπορούσε να είχε αλλάξει την συμπεριφορά της. Μόλις είδε δηλαδή ότι δεν υπήρχε περίπτωση να παραδοθεί η Ουκρανία. Είπατε για αυτή την ε, μετατροπή σε υπερνηστερία της Ουκρανίας. Ναι, είναι, είναι ένας κίνδυνος αυτός, αλλά όπως ε, ξέρετε και στο, στο γεύμα των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέθηκε το ίδιο θέμα. Αν θεωρούμε ότι υπάρχει ε, κίνδυνος η χώρα μας να μετατραπεί, να σε υπερνηστερία. Βλέπουμε αυτό βλέπουμε ότι οι Ρώσοι χρησιμοποιούν ξανά και ξανά αυτό το ίδιο υπόδειγμα. Χρησιμοποιούν, δηλαδή δημιουργούν μικρούς θύλακες, ε, τους παίρνουν με το μέρος τους, τους κατακτούν και στη συνέχεια προσπαθούν να δημιουργήσουν ε, υποτιθέμενες ε, δημοκρατίες ε, οι οποίες δεν, δεν μπορούν ποτέ να απεγκλωβιστούν από, τον, ε, ε από τον σφιχτό εναγκαλισμό με τη, με τη Ρωσία όπως έκαναν μόνο οι βαλτικές αυτή την πολιτική της Ρωσίας, της Ρωσίας πληρώνουμε με τη ζωή μας. Καταπολέμηση διαφοράς, αποκέντρωση. Εμείς διδασκόμαστε από άλλες χώρες της Ευρώπης, της Ανατολικής Ευρώπης, ιδίως από την Πολωνία, όταν προσπάθησε να ολοκληρώσει με τέτοια διαδικασία η Πολωνία για 9 χρόνια, όταν ε, αποφάσισε πλέον να γίνει συγχώνευση δήμων και κοινοτήτων ε, εμείς μια παρόμοια διαδικασία έχουμε διέλθει ε, δύο με τρία χρόνια ε, προσπαθούμε να πείσουμε ε, τους Δήμους και τις κοινότητες και τις περιφέρειές μας ότι θα τις, ε, θα τις ωφελήσει, θα έχουν περισσότερα χρώματα, περισσότερες αρμοδιότητες. Δεν έχουμε επίση όλες τις περιφέρειες ακόμη. Πώς σκοπεύουμε να ολοκληρώσουμε την αποκέντρωση και την συγχώνευση των δήμων και κοινοτήτων. Με κίνητρα ή θα γίνει απλά η διοικητική μεταρρύθμιση και θα επιβληθεί από τα πάνω για να δημιουργηθεί η νέα Ουκρανία. Αυτό προσπαθούμε όμως να κάνουμε στην, στην Ανατολική Ουκρανία προσπαθούμε να πούμε στους ανθρώπους εκεί ότι αυτά που θέλετε, τα δικαιώματα, όπως για παράδειγμα το να μιλάτε τη γλώσσα σας, μπορείτε να το επιτύχετε μέσω της αποκέντρωσης. Ήδη η νομοθεσία μας ε, προβλέπει ότι όλα τα έγγραφα πρέπει να μπορούν να συντάσσονται ε, και ε, στη γλώσσα της επιλογής τους. Μπορούν να καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει καταγραφεί αυτό κάπου ε, επίσημα σε νομοθεσία, αλλά ξέρετε, εμείς ε, στο κομμουνιστικό παρελθόν μας ακριβώς έχουμε τραύματα από την στάση των, ε, του κομμουνιστικού καθεστώτος απέναντι στην ουκρανική γλώσσα. Εγώ όταν ήμουνα ε, μαθητής έκανα δύο ώρες ε, την ε, εβδομάδα ουκρανικά στο σχολείο όπως και κάθε άλλη ξένη γλώσσα που διδασκόμασταν. Φαντάζεστε σε τι επίπεδο ήταν τα ουκρανικά μου όταν ήμουν παιδί. Οπότε περάσαμε μια διαδικασία ουκρανοποίησης της Ουκρανίας και κάποιες τοπικές κοινότητες βεβαίως δεν καταλαβαίνουν ίσως τη σημασία αυτής. Θέλω η ουγγρική μειονότητα να κατανοήσει ότι δεν μπορεί κανείς στα σοβαρά να περιμένει ότι ε, ε, σε σχολεία τα οποία χρηματοδοτούνται 100% από την οικονομική κυβέρνηση θα γίνεται διδασκαλία 100% ε, στα ουγγρικά. Θα υπάρξουν άλλες φόρμουλες για το πώς μπορούν να εντάσσονται τα μέλη αυτής της ουγγρικής εθνικής μειονότητας στο σχολικό σύστημα, πώς μπορεί να γίνει κανείς δικηγόρος, νομικός, ακόμη και διπλωμάτης. Θέλουμε λοιπόν να δώσουμε προτεραιότητα στην ουκρανική γλώσσα, στην ουκρανική ιστορία και βεβαίως να δοθεί και μια ισορροπία και κάθε εθνική μειονότητα να αποφασίσει τη δική της, ε, το δικό της μείγμα αν θέλετε, ποια θα είναι η δική της ισορροπία. Εμείς αυτή την ισορροπία επιδιώκουμε. Και αυτό που θέλουμε επίσης με τους Ούγκρους είναι, ε, συμφωνήσαμε ότι θα αναβάλουμε τον νόμο αυτό έως το 2023 αλλά οι Ούγγροι δεν βλέπω να ε, κοινοποιούν και να δημοσιεύουν και αυτοί ότι και εμείς κάτι κάνουμε. Είναι ένα θέμα που επανέρχεται ε, ξανά και ξανά όταν έχουμε επαφές με τους ε, διπλωμάτες ε, από την Ουγγαρία. Συναντήθηκα και με τον ομόλογό μου της Ουγγαρίας πριν από δύο εβδομάδες στη Νέα Υόρκη. Κανονίσαμε ότι θα γίνει και μια επίσκεψη του κυρίου Όρμπαν στην Ουκρανία. Δεν έχουμε βρει ακόμα ημερομηνίε. Έχουμε δύσκολο πρόγραμμα. Πάντω, σε κάθε περίπτωση, ε, σα είπα κιόλα ότι ό,τι και να προσπαθούμε να νομοθετήσουμε, έρχονται ομάδε ε, οι οποίε διαμαρτύρονται και διαδηλώνουν. Όσον αφορά την ιδιωτική τράπεζα στην οποία αναφερθήκατε, πρέπει και να ολοκληρώνω πάντως θα σας δώσω κάποιες εξηγήσει. Η ιδιωτική αυτή τράπεζα ήταν μεγαλύτερη τράπεζα μέχρι να ιδιωτικοποιηθεί. Και όπως λένε οι Αμερικάνοι θεωρεί το too big to fail, ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να καταρρεύσει η τράπεζα αυτή. Παρ' όλα αυτά άρχισε να μην τα πηγαίνει καλά και έπρεπε τότε να ληφθεί μία απόφαση που ενδεχομένω να μην ήταν πάρα πολύ δίκαιο προς τον τότε ιδιοκτήτη της αποφασίστηκε να ιδιωτικοποιηθεί εντελώ. Αυτό έγινε με απόλυτη διαφάνεια. Προσπαθούμε τώρα να το διερευνήσουμε περισσότερο. Αυτό δεν σημαίνει, και το έχει πει ο πρόεδρο Ζελένσκι, ότι η τράπεζα αυτή θα επαναθνικοποιηθεί. Δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο. Ο πρόεδρος Ζελένσκι το ξεκαθάρισε αυτό. Είπε ότι θα έπρεπε να διορθωθούν τα προβλήματα τα οποία έχει η τράπεζα αυτή. Θα πρέπει κατά ένα εντελώς ανεξάρτητο τρόπο να εξετάσουμε όλες τις εναλλακτικέ και η τράπεζα αυτή θα πρέπει να εξακολουθεί, όπως και στο παρελθόν που ήταν καθαρά δημόσια τράπεζα, να εξυπηρετεί τους Ουκρανούς πολίτες. Τώρα, ξέρετε ότι στις τελευταίες επαφές που είχαμε με τον πρόεδρο Λουκασέγκο της Λευκορωσίας και στις τελευταίες επαφές που είχε ο πρόεδρος Ζελένσκι με τον πρόεδρο Λουκασέγκο, συντοποιούν όλο και περισσότερο οι Ρώσοι θα έλεγα ότι αυξάνεται η πίεση απέναντί τους. Συντοποιούν τώρα και οι Λευκορώσοι ότι οι Ρώσοι δεν επικίνδυνοι μόνο για την Ουκρανία αλλά και για τη Λευκορωσία. Θα έλεγα ότι όλη η περιφέρεια το συντοποιεί τώρα αυτό και θα πρέπει οι Ρώσοι να το λάβουν αυτό υπόψη τους το καθεστώς του Πούτιν προσπαθεί να έχει όλο και μεγαλύτερη επιρροή και στη κυβέρνηση της Λευκορωσίας και στην επικράτηση της Λευκορωσίας και ως προς αυτό θα αντιδράσει η Λευκορωσία. Γι' αυτό το λόγο ο Λουκασέγκο δεν αποκαλεί πλέον τον εαυτό του ο τελευταίο ε, δικτάτορα. Αν δεν κάνω λάθο, τον τίτλο αυτό τον έχει δώσει στον Πούτιν. Είναι πάντω ένα ηγέτη ο οποίο βρίσκεται όλο και πιο κοντά στην Ουκρανία και στρέφεται όλο και περισσότερο προ την Ευρώπη. Συζητήσαμε μαζί του πολλά οικονομικά ζητήματα, μελλοντικά προγράμματα και έργα τα οποία θα θέλαμε να ελοποιήσουμε, τα οποία θα μα επιτρέψουμε να είμαστε πιο ενωμένοι για παράδειγμα να καταφέρουν να συνδυάσουμε περισσότερες οδούς μεταφορών προϊόντων, εσωτερικές πρωτες οδούς κτλ. Θα πρέπει να ολοκληρώσετε, λέει ο Πρόεδρος, τα επόμενα πέντε λεπτά. Σχεδόν ολοκλήρωσα, κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση των γεών. Δεν πρόκειται εδώ πέρα να σας πω ότι έχω πλήρη γνώση του ζητήματος αυτού. Η τελευταία μεταρρύθμιση περιλάμβανε 12-15 περίπου διαφορετικούς τρόπους ιδιωτικοποίησης. Αυτή τη στιγμή που, από όσο γνωρίζω, είμαστε από τις λίγες χώρες στον κόσμο που δεν επιτρέπουν άνευ περιορισμών την απόκτηση γης από ιδιώτες. Υπάρχουν συγκεκριμένε προϋποθέσεις που θα αποτρέψουν από καρτέλ να σφετεριστούν τα εδάφη της Ουκρανίας. Αυτό το οποίο προβλέπεται λοιπόν είναι ότι μόνο Ουκρανοί υπήκοοι θα μπορούν να αγοράσουν τις γης αυτές με συγκεκριμένες μόνο εξαιρεσει για συγκεκριμένους ξένους επενδυτές. Πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε περισσότερους επενδυτές για τα ουκρανικά εδάφη. Θα πρέπει να δούμε και συγκεκριμένε τεχνικέ λεπτομέρειε, πόσε εκτάσει μπορεί να κατέχει να αγοράσει ένα ξένο ιδιωτικό επενδυτή κ.ο.κ. Επίσης, ας μην ξεχνάμε ότι η τελευταία αυτή νομοθεσία εγκρίθηκε πριν από 11 χρόνια. Εκτοτε ανανεώνουμε εμείς το μορατόριο και θέλουμε ή δυνατόν το νέο αυτό εργαλείο να αρχίσει να χρησιμοποιείται στα πλαίσια του οικονομικού μας συστήματος. Και αναφέρομαι στη δυνατότητα δηλαδή πώληση και ιδιωτικοποίηση ενός τμήματος της εδαφικής επικράτειας της Ουκρανίας. Θέλουμε να ανοίξουμε λοιπόν την αγορά, αυτό προβλέπουμε από τον επόμενο Οκτώβριο και ο Υπουργό Οικονομικών μα προσπαθεί να δει ποια είναι τα οικονομικά μέσα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για να δοθούν δάνεια ή ακόμα και δυνατότητε μικροχρηματοδότηση σε πολίτες οι οποίοι θα θέλουν να αγοράσουν γη για να την εκμεταλλευτούν και που δεν έχουν του απαραίτητου πόρου. Δεν διατείνουμε ότι είμαι εδώ πέρα οικονομολόγο, προσπαθώντα με ένα πολύ σχηματικό τρόπο να σα εξηγήσω ποια είναι η προσέγγιση τη Ουκρανική κυβέρνηση σε σχέση με, το, με την μεταρρύθμιση αυτή που έχει να κάνει με τις ΓΕΣΕ. Τώρα όσον αφορά την ανταλλαγή κρατουμένων, όπως είπα πριν από λίγο, το ζήτημα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο για την Ουκρανία και θα έλεγα ότι θα έπρεπε εδώ πέρα να μιλάμε για μια παράλληλη ταυτόχρονη απελευθέρωση. Περί αυτού πρόκειται. Η επόμενη ανταλλαγή θα πρέπει να αφορά πάνω από 100 ανθρώπους. Και όντως ε, αυτή τη στιγμή έχουμε όλο και λιγότερους Ρώσους υπηκόους στις Ουκρανικές φυλακές, ενώ υπάρχουν πολύ περισσότεροι από την ρωσική πλευρά. Έχουμε Ρώσους φυλακισμένους, Ουκρανούς φυλακισμένους που βρίσκονται στη Ρωσία, άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στην κατεχόμενη Κρυμαία ή στα κατεχόμενα ανατολικά εδάφη της Ουκρανίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η εικόνα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και μπορείτε να καταλήξετε και εσείς τα δικά σας συμπεράσματα για το πόσο είναι εφικτό να ευοδοθεί αυτή η ανταλλαγή κρατουμένων. Ολοκληρώνω στο σημείο αυτό κύριε Πρόεδρε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα. Όντως οι προηγούμενες κυβερνήσεις την απαγόρευσαν την ύπαρξη του κομμουνιστικού κόμματος και δεν υπάρχουν πάρα πολλοί Ουκρανοί που έχουν μετανιώσει γι' αυτό. Ας μην ε, ξεχνάμε ότι το κομμουνιστικό καθεστώς ήταν αυτό το οποίο μας ε, έφερε σε κατάσταση εξαθλίωσης και δεν θα θέλαμε ουσιαστικά να επαναλάβουμε το πείρεμα αυτό. Από θεωρητικής πλευράς σας καταλαβαίνω, καμία ιδεολογία δεν θα πρέπει να απαγορεύεται. Αλλά στο παρελθόν ήταν το μόνο, το μοναδικό κόμμα, η μοναδική επιτρεπόμενη ιδεολογία. Εμείς ε, θεωρούμε ότι πολλοί από τους κομμουνιστές αυτές έχουν, έχουν γίνει τώρα σοσιαλιστές και ως Ουκρανική κοινωνία θεωρούμε ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο διαλλακτικοί και ανεκτικοί. Και νομίζω ότι ε, από θεωρητικής πλευράς τουλάχιστον καταλαβαίνω αυτό το οποίο ρωτήσατε. Δεν προβλέπουμε άμεσα μια κάποια αλλαγή. Μπορεί ενδεχομένως στο μέλλον να τροποποιηθούν κάπως τα πράγματα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε που αφιερώσετε τόσο χρόνο σήμερα μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε τόσο γρήγορα από το Λουξεμβούργο στις Βρυξέλλες. Σας ευχαριστούμε για όλες αυτές τις πληροφορίες που μας δώσετε και ευχόμαστε στη χώρα σας κάθε δυνατή θετική εξέλιξη. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε και το σημείο 11 διάφορα. Δεν θέλει να θίξει κανεί τίποτα στο σημείο αυτό. Η επόμενη συνεδρίαση θα λάβει χώρα στι 6 και 7 Νοεμβρίου εδώ στι Βρυξέλλε.